Μεγαλειότατε, εξ ονόματο όλων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήθελα να σα καλωσορίσω στο Στρασβούργο, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι μια μεγάλη τιμή για μα. Η παρουσία σα για τρίτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα και με τον τρόπο αυτό καταδεικνύεται το πνεύμα φιλίας και εμπιστοσύνης που σας διακατέχει έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ε, σήμερα βρισκόμαστε μέσα σε ένα έτος το οποίο έχει ξεκινήσει με πολλές ελπίδες, με την ελπίδα μιας δημοκρατικής άνοιξης, η οποία θα οδηγήσει σε ελευθερία έκφρασης, κράτος δικαίου και δημοκρατίας. Αυτό είναι και ο οικουμενικός πόθος των λαών της περιοχής σας. Εσείς έχετε με τις αποφάσεις σας καταδείξει την σοφροσύνη τη σοφροσύνη σας ως ηγέτη της Ιορδανίας έχετε λάβει αποφάσεις σόφρονες για μεταρρυθμίσεις στη χώρα σας και εμείς ως Ευρωπαίοι κοινοβουλευτικοί θέλουμε να υποστηρίξουμε την Ιορδανική κοινωνία σε αυτήν την πορεία μετασχηματισμού. Θέλουμε να σας βοηθήσουμε και στις σημαντικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις αλλά και στο πολιτικό άνοιγμα της χώρας σας. Έχετε την απόλυτη υποστήριξή μας. Στις 12 Ιουνίου 2011, στον λόγο που εκφωνήσατε ενώπιον του Ιρδανικού λαού, τονίσατε ότι είσαστε έτοιμος να προχωρήσετε σε εκλογές κοινοβουλευτικές και με την συμμετοχή ε, όλων να μπορέσει να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Και στη συνέχεια να λειτουργήσετε επί τη βάση μιας κοινοβουλευτική πλειοψηφία επί της οποία θα οικοδομηθεί μια κυβέρνηση στην Ιορδανία. Εμείς χαιρετίζουμε τη σαφήνεια της έκφρασης αυτών των βασικών αρχών και της αποδοχής του κράτους δικαίου και της δημοκρατικής λειτουργίας ενό κράτους. Εμείς, από την άλλη πλευρά, θέλουμε να τονίσουμε ότι είναι απαραίτητο να αντιδράσουμε στην βία την τρομοκρατία και την απογοήτευση που πολλές φορές δημιουργείται στους πολίτες. Με το δικό σας τρόπο εσείς έχετε αποτρέψει αυτό για τους πολίτες της Ιορδανίας και έχετε δείξει ένα διαφορετικό δρόμο. Εμείς σας υποστηρίζουμε σαν φίλοι και σαν εταίροι και είμαστε διατεθειμένοι να σας υποστηρίξουμε απόλυτα να μπορέσετε να φέρετε σε πέρας τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες έχετε υποσχεθεί για την Ευρώπη. Η Ιορδανία είναι μια χώρα με την οποία βρισκόμαστε σε δεσμούς βαθιάς φιλίας και υπογραμμίζω και τη δική σας προσωπική δέσμευση <clears throat> που φάνηκε τις τελευταίες εβδομάδες ήδη με την πρότασή σας να διαμεσολαβήσετε μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων ώστε να μπορέσουν να επανέλθουν και οι δύο πλευρές στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων. Όλα αυτά μας δείχνουν ότι είσαστε ένα σύμμαχό σας στον αγώνα για τη δημοκρατία και την ειρήνη στη Μέση Ανατολή και <clears throat> επίσης για την ελευθερία. Μεγαλειότατε, με μεγάλη χαρά σας δίνω τον λόγο. Στο όνομα του Θεού, του Φιλές Φλαχνού, του Ελεήμονος, κύριε Πρόεδρε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας ευχαριστώ όλους σας για τη θερμή σας υποδοχή. Οι δεσμοί μεταξύ της Ιορδανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ στερεοί. Είναι κάτι που βρίσκεται στο κοινό μας συμφέρον να υπάρξει ευμάρεια και σταθερότητα σε όλη την περιοχή μας, σε όλη τη γειτονιά μας. Και είναι κοινή πεποίθησή μας ότι πρέπει να έχουμε μια τέτοια σχέση γειτονίας. Μια σχέση γειτονίας την οποία αξίζουν και οι λαοί μας. Η οποία να χαρακτηρίζεται από ελευθερία και ανθρώπινη αξιοπρέπεια και να δίνει τη δυνατότητα και την ευκαιρία της προόδου μέσα στη σταθερότητα και την ειρήνη. Όταν μιλάω για την γειτονία μας και το μέλλον της περιοχής μας. Αυτό είναι ένα εγχείρημα κοινό και γι' αυτό θέλω να λάβω το λόγο σήμερα. Ξεδιπλώνεται η αραβική άνοιξη στον κόσμο μας. Δεν πρόκειται να κρατήσει μονάχα το χρονικό διάστημα μιας εποχής, ενός τριμήνου, ούτε καν ενός έτους. Οι κοινωνίες μας αντιμετωπίζουν την πρόκληση του να περάσουν από τη διαμαρτυρία σε προγράμματα και δράση, από τις επικρίσεις σε οικοδόμηση εθνικών στρατηγικών. Η κάθε χώρα θα ακολουθήσει το δικό της δρόμο. Θα είναι διαφορετική αυτή η δρόμη. Κάποιες χώρες συζητούν με προσπάθεια επίτευξης συνένεσης. Αλλού όμως βλέπουμε να υπάρχει διχόνοια και αντίδραση που προκαλεί αστάθεια, βία και αυτό έχει επιπτώσει και σε περιφερειακό επίπεδο. Υπάρχουν και εξωτερικοί παράγοντες οι οποίοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτή την αστάθεια και αυτές τις διχόνοιες. Υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι, μεγάλες αβεβαιότητες που είναι πραγματικές. Αλλά θέλω να εκφράσω την άποψη εκατομμυρίων ανθρώπων όταν λέω ότι ο αραβικός κόσμος έχει ξυπνήσει και είναι έτοιμος να αδράξει τις προκλήσεις που έχει ενώπιον του. Αυτοί οι οποίοι ήθελαν να δουν τα μηνύματα αυτής της αλλαγής τα είχαν δει ήδη από το παρελθόν. Για δεκαετίες οι άνθρωποι της περιοχής του αραβικού κόσμου θέταν ερωτήματα, είχαν προσδοκίες, θέλαν να βρουν μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα είχαν νόημα και θέλαν να ενισχυθεί η κοινωνία των πολιτών, ιδίως να αυξηθεί ο ρόλος των γυναικών και επίσης των νέων που τώρα συνδέονται με ένα παγκόσμιο πλέγμα ψηφιακής επικοινωνίας. Οι παγκόσμιες κρίσεις στα χρηματοπιστωτικά, τα προβλήματα στην αγορά ενεργείας. Όλα αυτά έχουν πλήξει τις οικονομίες μας. Οι οικογένειες που έχουν θυσιάσει πολλά για να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους βλέπουν τα νέα παιδιά τους να έχουν προετοιμαστεί για θέσεις εργασίας που δεν υπάρχουν καθόλου. <clears throat> Σήμερα η περιοχή στην οποία ζω αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη αργία των νέων οποιοδήποτε τμήματος του κόσμου. Είπανε κάποιοι ότι αυτό είναι η απώλεια μιας γενιάς. Είναι κάτι που αφορά εκατό εκατομμύρια νέων. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα νέων στην ιστορία μας που βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση. Ξέρω ότι αυτό σας ενδιαφέρει και σας απασχολεί και εσάς στην Ευρώπη. Είναι το ίδιο πρόβλημα. Οι περιοχές μας έχουν διαφορετική δημογραφική πυραμίδα και εξέλιξη. Αλλά έχουν κοινά προβλήματα και κοινέ ανησυχίες. Οι νέοι της, σήμερα είναι το μέλλον της αύριον. Δεν μπορούμε να αφήσουμε ούτε ένα νέο να βρεθεί σε κατάσταση απόγνωσης χωρίς θέση απασχόλησης. Αυτή η πραγματικότητα είναι αυτή που κατευθύνει τις προσπάθειες της Ιορδανίας. Εμείς θεωρήσαμε ότι αποτελεί και μια ευκαιρία. Θεωρούμε ότι είναι μια ευκαιρία να ξεπεράσουμε τα προσκόμματα του παρελθόντος, να έχουμε μια μεταρρύθμιση η οποία θα αποδώσει καρπούς. Πέρσι κάναμε κάποια άμεσα βήματα για να προχωρήσουμε σε εθνικό διάλογο, για να οικοδομήσουμε τη συνένεση επί τη βάση συγκεκριμένων δράσεων και σχεδίων. Και καταρχήν εστιάσαμε στη διαμόρφωση ενός συντάγματος που είναι το θεμέλιο των πολιτικών συστημάτων. Τον προηγούμενο Σεπτέμβρη, μετά από τις συστάσεις μιας Εθνικής Επιτροπής, το 1 τρίτο του συντάγματος έγινε δεκτό. Έχει νέες διατάξεις με ευρύτερη εκπροσώπηση, ενίσχυση των, των πολιτικών κομμάτων, προστασία των ε, ε, αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων και διαχωρισμό εξουσιών. Επίσης υπάρχει νέα νομοθεσία για τα πολιτικά κόμματα και για τις εκλογές. Συγχρόνως έχει εγκριθεί νομοθεσία για το νέο συνταγματικό δικαστήριο και για την Ανεξάρτητη Εκλογική Επιτροπή στην Ιορδανία. Η επόμενη δοκιμασία μας θα είναι οι δημοτικές καθώς και οι βουλευτικές εκλογές. Ως εγγυητής της πολιτικής διαδικασίας μεταρρυθμίσεων έχω παροτρύνει και την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ορδανίας να τηρήσουν το θεσπιστέν χρονοδιάγραμμα και να εγκρίνουν το ταχύτερο δυνατόν τα βασικά στοιχεία της νέας νομοθεσίας, χωρίς όμως να θυσιάσουν τον περιεκτικό χαρακτήρα αυτής της διαδικασίας μεταρρύθμισης. Μόνο εμεί, οι Ιορδανοί, μπορούμε να οικοδομήσουμε το μέλλον τη Ιορδανία και θα πρέπει να το πράξουμε αυτό με τέτοιο τρόπο ώστε η χώρα μα θα παραμείνει μια ασφαλή χώρα, ένα ασφαλή λιμένας παρά τις ταραχές, παρά τι θύελε που ξεσπούν στην περιοχή μα παρά τι οικονομικέ και ενεργειακές κρίσεις που μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε μεταρρυθμίσεις που βασίζονται στη συνένεση, που βασίζονται σε διαρθρωτική πλήρη αλλαγή στον πολιτικό, τον οικονομικό και τον κοινωνικό στίβο. Πάντα με σεβασμό των δικαιωμάτων και των ελευθεριών όλων των πολιτών μας. Στη διαδικασία αυτή η Ιορδανία μπορεί να αποστεί ένα παράδειγμα για όλες τις χώρες της περιοχής ό,τι αφορά τη δημοκρατική εξέλιξη και τη μεταρρύθμιση. Είμαι απόλυτα πεπισμένο ότι το 2012 θα είναι ένα κομβικό έτος σε σχέση με τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις στην Ιορδανία. Μεταξύ των πιο σημαντικών μέτρων είναι η οικοδόμηση μιας ισχυρής και ανθεκτικής κομματικής δομής και πολιτικής και κοινοβουλευτική δομής στην Ιορδανία. Ξέρουμε ότι αυτό δεν αφορά μόνο την τωρινή πολιτική τάξη αλλά και τις επερχόμενες ε, γενιές πολιτικών. Με τον τρόπο αυτό θα δείξουμε ότι λειτουργεί το πολιτικό σύστημα στην Ιορδανία. Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα και εκτιμούμε ιδιαίτερα την αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτών των μεταρρυθμίσεων. Πριν από δύο μήνες η ειδική μονάδα Ευρωπαϊκή Ένωση Ιορδανία συναντήθηκε για να συζητήσει τα κέρια προγράμματα τα οποία υποστηρίξουν τι προτεραιότητέ μα στον τομέα των μεταρρυθμίσεων. Δημοκρατικού θεσμού, κοινωνία των πολιτών, δημιουργία θέσεων απασχόληση. Όλα αυτά θα προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη και επίσης θα βοηθήσουν τους πολίτες μας να είναι ελεύθεροι. Έχουν περάσει, θα έχουν περάσει σύντομα 10 χρόνια από την έγκριση της Συμφωνίας Σύνδεσής μας. Αυτό άνοιξε ευκαιρίε και θέσει απασχόληση και από τι δύο πλευρέ τη συμφωνία. Ελπίζω ότι αυτέ οι ευκαιρίε, οι οποίε τώρα ενισχύονται από το αναβαθμισμένο επίπεδο εταιρική μα σχέση, θα ανθίσουν ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια η Ιορδανία ακολούθησε μια σειρά από εθνικούς στόχους παρά τις συγκρούσεις στην ευρύτερη περιφερειά της. Αγαπητοί μου φίλοι όμως, η ειρήνη θα πρέπει να εδρεωθεί για να μπορέσει να ανθίσει οικονομικά και να είναι ασφαλής η περιοχή μας. Δεν μπορούμε να έχουμε ακόμα μια γενιά η οποία θα περιμένει να λυθεί το πρόβλημα της Παλαιστίνης. Εδώ και δέκα χρόνια οι αραβικές χώρες όλες μαζί ζήτησαν να υπάρξει μια δίκαιη ειρήνη. Πήραμε την απόφαση σαν αραβικές χώρες να κοιτάξουμε προς το μέλλον, να γνωρίσουμε το παρελθόν, να αναζητήσουμε συμφωνία και να αποδεχθούμε και άλλες θέσεις. Η Αραβική Πρωτοβουλία για την Ειρήνη αναγνωρίστηκε από όλους όσους αγαπούν την ειρήνη στον κόσμο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα υπόλοιπα μέλη του λεγόμενου κουαρτέτου. Ζητάμε και από το Ισραήλ να εμπλακεί στην πρωτοβουλία αυτή. Η Αραβική Ειρηνευτική Πρωτοβουλία βασίζεται στη μοναδική δυνατή λύση. Δύο κράτη, το ένα πλάι στο άλλο, με αξιοπρέπεια, με αποφασιστικότητα, αυτοδιάθεση μια ανεξάρτητη βιώσιμη Παλαιστίνη στα σύνορα τα αναγνωρισμένα με την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσά της. And collective peace and security guarantees for Israel. Επίσης εγγυήσεις για το Ισραήλ. And a final settlement in accordance with σύμφωνα με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με το συμπεφωνισμένο ψήφισμα σχετικά με το τελικό καθεστώς. Η πρωτοβουλία αυτή θα διασφαλίσει την ειρήνη ανάμεσα στο Ισραήλ και τους Άραβες γείτονες και το δέχεται το σύνολο του αραβικού κόσμου. Προσφέρεται η λύση αυτή εδώ και δέκα χρόνια point to the change in the Arab world. Προβλέπεται μία λύση η οποία θα αλλάξει πολλά και στον αραβικό κόσμο και έτσι δείχνουμε ε, προς το Ισραήλ ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε πλέον. Δεν υπάρχει χρόνος. Η αραβική ίνιξη άνοιξη ξέρετε ότι βασίζεται σε μία έκκληση εκ βάθους για μια νέα προσπάθεια για την ειρήνη και να μην υπάρχουν πλέον προσβολές και η Ισραηλινή κατοχή είναι μια τέτοια η χειρότερη από όλες τις προσβολές. Συνεχίζονται οι επικισμοί, δημιουργούνται περισσότερες δυσφορίες, περισσότεροι κίνδυνοι και προβλήματα. Εάν κάνουμε αυτό το βήμα όπου δεν θα είναι πλέον εφικτή η λύση με δύο ανεξάρτητα κράτη, τότε το Ισραήλ θα είναι πραγματικά μακράν περισσότερο από ποτέ από την επιθυμητή ασφάλεια και θα χρειαστούν δύο γενιές τουλάχιστον για να υπάρξει μια νέα πρωτοβουλία για την ειρήνη. Εμείς θεωρούμε σαν Ιορδανία ότι μια τέτοια πορεία για την ειρήνη είναι ηθικό μας καθήκον αλλά είναι και προς το συμφέρον μας και συνεχίζουμε να την επιδιώκουμε. Στο Αμάν φέτος φέραμε σε επαφή επανειλημμένα τους διαπραγματευτές από τις δύο πλευρές. Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε χωρίς την τεράστια προσπάθεια που έκανε και η ευρωπαϊκή διπλωματία η ιδιαίτερα δραστήρια υποστήριξη της Ευρώπης η οποία συνέχισε να πιέζει όλους για την ειρήνη. Και έτσι η αελπίδα παραμένει ζωντανή. Πράγματι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ένας πολύτιμος φίλος και για τις δύο πλευρές, για αυτούς που εργάζονται για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Οι προκαταρκτικές αυτές συνομιλίες στο ΑΜΑΝ είναι ένα μικρό βήμα, δίνουν τη δυνατότητα στις δύο πλευρές να αποκαταστήσουν τις διμερείς επαφές και τώρα όμως η διαδικασία απαιτεί αν θέλετε ένα νέο ποιοτικό άλμα μια νέα εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Αραβικό κόσμο είναι κάτι το απαραίτητο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε τα πρώτα βήματα υπέρ της λύσης των δύο κρατών και κατά τη συνέχιση των επικισμών που δημιουργούν προσκόμματα στην πρόοδο της ειρηνευτικής διαδικασίας. Καταλαβαίνετε τους κινδύνους παγκόσμια που παρουσιάζει η σύγκρουση στην περιοχή και ε, φυσικά έχετε τεράστια αξιοπιστία λόγω των εμπειριών σας και λόγω της ε, εμπειρίας που έχετε στα πλαίσια της δημιουργίας δημοκρατικών θεσμών, σταθερότητας και εμπιστοσύνης. Η εμπειρία αυτή ελπίζω να σας είναι και σε εσά χρήσιμη τα επόμενα χρόνια. Αγαπητοί φίλοι, πολλοί λαοί, μία γειτονία όμως και ένα κοινό μέλλον για όλους. Αυτή είναι η πρόκληση και για την ειρήνη και την Ευρώπη και την Μέση Ανατολή. Αυτή είναι και η δική μας ισχύ. Μαζί θα αντιμετωπίσουμε τα τεράστια προβλήματα, είτε είναι οικονομικά είτε είναι πολιτικά. Μαζί θα αναζητήσουμε την ειρήνη. Οι λύσεις είναι περίπλοκες και ο δρόμος προς την ειρήνη είναι και αυτός πολύ δύσκολος, αλλά από κοινού έχουμε θα έλεγα την επιθυμία, τη βούληση και την σοφία που απαιτείται για να μπορέσουμε να πετύχουμε. Ευχαριστώ. Μεγαλειότατε, σας ευχαριστούμε για την ομιλία σας. Σας ευχαριστούμε για τα λόγια σας. Νομίζω ότι τα χειροκροτήματα των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταδεικνύουν ότι υπάρχει μια μεγάλη ομοφωνία μεταξύ ημών και ημών σε σχέση με τη διαδικασία αυτή και σε σχέση με το τι μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια και της συνεργασίας της Ιορδανίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και έναντι όλων των χωρών της ευρύτερης περιοχής σας. Νομίζω λοιπόν ότι όπως αναφέρθηκε και στα δικά σας λόγια η Ευρώπη έχει να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην διαμεσολάβηση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για τον λόγο σας και θέλω και πάλι να τονίσω ότι νομίζω ότι τα χειροκροτήματα τα οποία συνόδευσαν το τέλος του λόγου σας καταδεικνύουν ότι όλοι μας θέλουμε να υποστηρίξουμε μια στεναρή και ισχυρή πολιτική και οικονομική ανάπτυξη όχι μόνο στην Ιορδανία αλλά στο σύνολο της περιοχής ως υπόβαθρο για μια ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και προς Ανατολής. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν.